Äh, Καλησπέρα αγαπητοί συνάδελφοι. Ας αρχίσουμε τη σημερινή μας συνεδρίαση. Έχουμε λιγότερες γλώσσες σήμερα και έχουμε διερμηνία αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά και ελληνικά. Και έχουμε και εστονικά αλλά παθητικά μόνο. Έχετε την ημερήσια διάταξη και αν δεν έχετε κάποια παρατήρηση θεωρώ ότι εγκρίνεται η ημερήσια διάταξη. Στις ανακοινώσεις του Προέδρου θα ήθελα να σας πω ότι σιγά σιγά πλησιάζουμε στο τέλος των εργασιών μας. Και στα έγγραφα τεκμηρίωσης που προετοιμάζουμε θέλουμε να προετοιμάσουμε τι θα κάνουμε και θέλουμε να βάλουμε και μια φωτογραφία των μελών της Επιτροπής. Και γι' αυτό τη Δευτέρα, όταν θα κάνουμε την ψηφοφορία στην Επιτροπή, θα έχουμε και ένα φωτογράφο του Κοινοβουλίου. Σα το λέω για να προετοιμαστείτε, να γίνετε ωραίοι για την επόμενη Δευτέρα, για να βγείτε ωραίοι στη φωτογραφία. Και για να είναι και η έκθεσή μας πιο ευπαρουσίαστη. Στο τρίτο σημείο έχουμε την έγκριση των πρακτικών της, της συνεδρίας συγγνώμη, της 11 η Απριλίου, 12 Απριλίου και 5 η Μαΐου. Έχουν διανεμηθεί τα πρακτικά και θεωρώ ότι εγκρίνονται αφού δεν έχετε παρατηρήσεις. Και περνάμε στο κύριο σημείο που έχουμε για σήμερα. που είναι οι συμβιβαστικέ προτάσει, τι οποίε ελπίζουμε να ολοκληρώσουμε. Έχουμε ήδη κάνει αρκετέ συνεδριάσει ώστε από τις 600 τροπολογίες που είχε η να φτάσουμε τώρα στο τελικό κείμενο μετά τις συμβιβαστικές τροπολογίες της Πεβάνς. Έχουμε κείμενα μέσα σε πλαίσια όπου δεν έχουμε ολοκληρώσει τις εργασίες μας, δεν έχουμε φτάσει στο τελικό τελικό κείμενο, διότι εδώ κάποια μέλη έχουν ακόμη κάποιες τροπολογίες, χρειάζονται κάτι όπως χωριστή ψηφοφορία ή, εν πάση περιπτώσει, υπάρχει κάποια εκκρεμότητα για αυτά που είναι εντός πλαισίου. Και θα δώσω τώρα το λόγο στην Περβάνς που θα μας παρουσιάσει το κείμενο και τις εκκρεμότητες που παραμένουν. Θέλω να σας ζητήσω συγγνώμη, αλλά έχω σήμερα το απόγευμα μια συνάντηση στο Düsseldorf που δεν μπορούσα να την αναβάλω και γι' αυτό θα, πρέπει, να φύγω στις 4, θα πρέπει να φύγω ίσως ε, και νωρίτερα αλλά σας ζητώ συγγνώμη από τώρα. Περιβόνος, λοιπόν, έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ όλους τους ε, συναδέλφους, διότι πιστεύω ότι και ιδιαίτερα τους συντονιστές και τους σκιώδεις ε, εισηγητές, με τους οποίους νομίζω ότι τη Δευτέρα είχαμε μια συνάντηση εξαιρετικά χρήσιμη που εξελίχθη σε ένα πνεύμα συνεργάσιμο, πνεύμα συνεργασίας, όπου όλοι μπόρεσαν να παρουσιάσουν τις ε, προτάσεις τους και προσπάθησαν να πετύχουν μια σύγκληση προς επίτευξη συμφωνίας. Όπως είπατε, απομένουν κάποια σημεία. Πάνω σε αυτά Θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε την ευκαιρία αυτής της συζητήσεως για να τελειοποιήσουμε κάποιες πτυχές. Πριν το κάνουμε αυτό, θα ήθελα απλώς να θέσω το πλαίσιο. Να σας πω ε, για τη συνεδρίαση που αφορά το Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση. και ασχοληθήκαμε με την χρήση, την κινητοποίηση αυτού του ταμείου. Είχαμε να εξετάσουμε δύο περιπτώσεις και αφορούσαν τη Δανία. Όπως φαντάζεστε, είναι από τις χώρες μοντέλα της Ευρώπης ε, από πολλές πλευρές. Όμως, οι δύο υποθέσεις που εξετάσαμε αφορούσαν η μία το κλείσιμο ενός ναυπηγείου που είχε πάρα πολύ καλές επιδόσεις, πάρα πολύ σύγχρονο ναυπηγείο που μειώνει τις δραστηριότητες του για να ανοίξει στην Ασία. Και άλλη περίπτωση, μία ένα εργοστάσιο κατασκευής ε, μονάδων παραγωγής από ηλική ενέργεια που μειώνει την παραγωγή για να ανοίξει μονάδες παραγωγής στην Ασία, λέγοντας ότι πρέπει να είναι πιο κοντά στα κέντρα τελικής κατανάλωσης. Γιατί τα λέω αυτά. Δεν λέω για να δώσω δραματικό τόνο στη συζήτησή μας, αλλά κάτι δείχνει αυτό. Σε σχέση με τους ανατολισμούς που ακολουθήσαμε στην πρώτη προσωρινή ενδιάμεση έκθεση, όπου είπαμε ότι πρέπει να δούμε από πού μπορούμε να ξαναδημιουργήσουμε τη η αξία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και βλέπουμε πόσο δύσκολο είναι το έργο που έχουμε μπροστά μας. Οι προτάσεις που θα κάνουμε ε, θα συμβάλλουν στη βελτίωση της καταστάσεως, όμως είναι τεράστια ακόμα η πρόκληση που έχουμε μπροστά μας. Πέρα από τα παραδείγματα που σας ανέφερα. Στο κείμενο που σας υπευλήθη, Σας προτείνω να εξετάσετε λεπτομερέστερα τα κουτάκια, αν θέλετε, εκεί, στα πλαίσια αυτά, τα πλαισιωμένα κομμάτια που ίσως εκεί ε, τονίζονται τα εκκρεμούντα προβλήματα. Πριν να το κάνουμε αυτό, να σε πιστήσω την προσοχή στην αιτιολογική σκέψη προτείνω να θεθεί στο κείμενο το συμβιβαστικό, διότι ανέλαβα υποχρέωση έναντι των συντονιστών και των σκιωδών εισηγητών στη συνεδρίασή μας, δεσμεύτηκα να προτείνω ένα κείμενο που θα μας επιτρέψει να αναφερθούμε στα διακυβευόμενα όσον αφορά την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων που ίσως υπονομεύεται το όλο καθεστώς όπως ξέρετε σήμερα έχει γίνει εύθραυστο. Έχει γίνει εύθραυστο θέμα της ελευθερής κυκλοφορίας. Λοιπόν, έχω ένα κείμενο μια αιτιολογικής σκέψη που προτείνω να προσθεθεί και θα ήθελα να ακούσω ποια είναι τα σχόλια των συναδέλφων όσον αφορά αυτή την ενδεχόμενη προσθήκη. Όσον αφορά την παράγραφο 17α, νέα, διότι είναι η πρώτη παράγραφος η οποία εξακολουθεί να παρουσιάζει προβλήματα. Εκεί θα ζητηθεί ξεχωριστή ψηφοφορία, αυτό πιστεύω, όσον αφορά το τελευταίο τμήμα της φράσης, αλλά θεώρησα ότι στη συμφωνία που συζητήσαμε, εν πάση περιπτώσει και στο τελευταίο τμήμα της φράσης, ο όρος σε τρίτες χώρες δεν εμφανιζόταν. Άρα η ξεχωριστή ψηφοφορία θα πρέπει να είναι καλή για τη διάλυση, των, την άρση των εμπορικών φραγμών, χωρίς όμως σε τρίτες χώρες, χωρίς την αναφορά το κομμάτι που λέει σε τρίτες χώρες. Ε, στην παράγραφο 19 οι πράσινοι νομίζω ζητούν ξεχωριστή ψηφοφορία όσον αφορά τη λέξη fully Η λέξη free, δηλαδή αναφορά στην δίκαιη και ελεύθερη, στο δίκαιο και ελεύθερο εμπόριο, όσον αφορά τη λέξη free, ελεύθερο. Στην παράγραφο 21, ίσως ζητηθεί ξεχωριστή ψηφοφορία από το ΕΛΚ που ενισχύει για κάτι που επελήθη στην τελευταία εκδοχή κατά την άποψή μου της τροπολογίας αλλά θα πρέπει να το εξακριβώσουμε αν ισχύει και μετά ε, και το EFD όπως αναφέρεται στον κατάλογο δεν θα υποστηρίξει αυτή την παράγραφο. Συγγνώμη που σε διακόπτω λέει ο πρόεδρος, ο πρόεδρος. Υπάρχει ένα προβληματάκι γλωσσικό transformed into a world economic council, ότι μεταμορφώνεται το into. Αντί in να γίνει into στα αγγλικά. Μεταμορφώνεται εις ένα συμβούλιο οικονομικό κλπ. Το into αντί το in. Δεν έπρεπε να λέει in αλλά into. Η κυρία Περέζη είναι εκτός μικροφώνου γιατί την ακούμε. Λοιπόν, στην παράγραφο 27 σε λατινικό νέο Ζητείτε ξεχωριστή ψηφοφορία και οι πράσινοι το ζητούν και οι σοσιαλιστές και οι δημοκράτες για το τελευταίο κομμάτι του κειμένου διότι δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε το αίτημα μιας ανάπτυξης μιας Ευρώπης των ε, υπηρεσιών και διεύρυνση, αύξηση του εμπορίου σε αυτό το τομέα. Στην παράγραφο 29D λατινικό, νέο, εδώ γίνεται αναφορά στις δημόσιες υπηρεσίες και κατά πόσο θα πρέπει απλώς να ζητηθεί η διατήρηση των δημοσίων υπηρεσιών στην περίοδο λιτότητας και περιορισμών που, στην οποία βρισκόμαστε ή αν αυτή η μέρημνα, αυτή η ανησυχία για το μέλλον των δημοσίων υπηρεσιών αφορά μόνο αυτές που είναι οι ουσιαστικές. Εξού και το αίτημα ξεχωριστής ψηφοφορίας όσον αφορά τον όρο ουσιαστικές. Essential. Όσον αφορά το εδάφιο 4 της παραγράφου 34 η ομάδα ECR έχει πρόβλημα αλλά νομίζω ότι θα μπορούσαν να εξηγήσουν πού έγκυται το πρόβλημά τους, τι τους δημιουργεί το πρόβλημα. Στην παράγραφο 37 Εδώ πρόκειται περί δυσκολίας που αντιμετωπίζει η EFD, η ομάδα, και για την 37 και για την 37α νέα. Όσον αφορά την 38, τη συμβαστική για την παράγραφο 38, το ΕΛΚ ζήτησε ξεχωριστή ψηφοφορία όσον αφορά τις, τη συγχώνευση των δικτύων ε, των ε, ε, χρηματιστηρίων. Δεν είναι θέμα συγχωνεύσεων, λέει ο Πρόεδρος. Για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, δηλαδή εκπλήττομαι για το αίτημα αυτό η ξεχωριστή ψηφοφορία από το ΕΛΚ. Διότι όπως είπα και στις διαπραγματεύσεις, οι χώρες θέλουν να ευνοήσουν την προσέγγιση, την πρόσβαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην αγορά. Και θεωρείται ότι έτσι οδηγούμεθα σε μια ποικιλομορφία της ε, χρηματοδότησης των επιχειρήσεων. Και ότι υπάρχει πρόσβαση σε περισσότερες πηγές χρηματοδότησης όταν αυτό είναι πρόβλημα τώρα, η χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και οι πηγέ χρηματοδότηση αυτών, γιατί να μην υποστηριχθεί μια τέτοια πρωτοβουλία, εφόσον πρόκειται περί ρυθμισμένων αγορών, πολύ καλά ρυθμιζομένων αγορών, που λαμβάνουν υπόψη τους στόχους της σταθερότητας και της βιωσιμότητας. Όσον αφορά την παράγραφο 41, αφορά τα θέματα τα φορολογικά, και εδώ έχει υπάρξει αίτημα για ξεχωριστή ψηφοφορία, διότι έχουμε διαφωνία όσον αφορά την φύση της φορολογητέας βάσης. Τι εννοούμε όσον αφορά την ενοποιημένη βάση φορολόγησης των επιχειρήσεων. Κάποιοι αρκούνται ε, στην πρόταση δυνητικής, την εθελοντική που παρουσίασε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και άλλοι θέλουν αυτή η ενοποιημένη φορολογητέα βάση να είναι υποχρεωτικής φύσεως, που εγώ θεωρώ ότι είναι η μόνη δυνατή βάση, αν θέλουμε να προχωρήσουμε σε αυτόν τον τομέα και να αποφύγουμε να υποβάλουμε μια πρόταση η οποία θα είναι μια πρόταση ε, σε, κατά παραγγελία των πολυεθνικών που θέλουν να μεγιστοποιήσουν να μειώσουν στο να μεγαλιστοποιήσουν τα κέρδη τους πάνω Όσον αφορά την τροπολογία 43, συμβαστική τροπολογία, η ομάδα του ΕΛΚ δεν ήθελε να υποστηρίξει αυτή την παράγραφο. Είμαι έτοιμη να το ξανασυζητήσω. Αλλά μια έκθεση αυτή έχει το πλεονέκτημα να μπορεί να θέτει αυτά τα ερωτήματα. Όσον αφορά την παράγραφο 43, εδάφιο 3, υπάρχει έτοιμα ξεχωριστή ψηφοφορία από πλευρά DFD και όσον αφορά την παράγραφο 44α νέο και 44β νέο μισό λεπτό Δεν υπάρχουν προβλήματα, δεν υπάρχει καμία δυσκολία σε αυτό το κείμενο. Απλώς το κείμενο αρχικά συγχωνεύτηκε, συμφώνησαν συντονιστές να παρουσιαστούν δύο ξεχωριστές παραγράφοι. Μου λέει κάποια ομάδα ότι έχει κάποια δυσκολία, αλλά δεν το κουβεντιάσαμε ακόμα. Για την παράγραφο 45, η ομάδα ECR θα εκφράσει τη θέση της για την παράγραφο 46 που αφορά την ευέλικτη ασφάλεια, flexi security. Οι πράσινοι είπαν ότι ε, δεν, έχουν, δεν είναι πολύ πρόθυμοι να υποστηρίξουν την πρόταση. Εγώ θα ήθελα, εν πάση περιπτώσει, σε αυτή την παράγραφο να διεξαχθεί ξεχωριστή ψηφοφορία όσον αφορά τη μη σωστή εφαρμογή τη ευέλικτη ασφάλεια improper implementation of Lexi Security, ούτως ώστε να μπορέσουν να τοποθετηθούν όσοι ενδιαφέρονται για αυτό το θέμα. Στην παράγραφο 50, η ομάδα του ECR και του EFT είχαν πρόβλημα να στηρίξουν τη συμβιβαστική λύση, όπως και η EFT δεν υποστηρίζει την παράγραφο 50, όπως βλέπετε την 50α, η ευθύνη υποστηρίζει την 50α, ούτε την συμβιβαστική για την παράγραφο 51, ούτε η ομάδα του ECR την υποστηρίζει. Το ίδιο ισχύει όσον αφορά το ECR για την παράγραφο 51b, λατινικό, που είναι μια παράγραφος που ζητά μια ισχυρή Ευρωπαϊκή Επιτροπή, παράγραφος 52 τη συμβαστική 52. Δεν την υποστηρίζει ούτε το ECR, ούτε το EFT. Είναι παράγραφος που απευθύνει μια έκκληση υπέρ της κοινοτική μεθόδου και συμπεριλαμβανομένης σημαντικής συμμετοχής των Εθνικών Κοινοβουλίων, παράγραφος 56. Και εδώ υπάρχει αίτημα για μια Ευρώπη της σύγκλησης και της αλληλεγγύης που απαιτεί μεγαλύτερη συνοχή δαπανών και αρμοδιοτήτων σε ευρωπαϊκή κλίμακα δεν έπρεπε να βάλουμε δαπάνε spending γιατί αν λέμε δαπάνε spending σημαίνει και μέσα, means. Άρα πρέπει να λέμε budget πρέπει να κάνω προφορική τροπολογία όσον αφορά τη λέξη spending, τις δαπάνες. Δεν μπορούμε να κάνουμε μόνο αυτό, να δαπανούμε. Χρειάζονται και άλλα μέσα, means. Όσον αφορά τη συμβαστική 57, δεν την υποστηρίζει η EFD. Είναι μια παράγραφος ε, σημαντική, παρουσιάζει ένα όραμα. Είναι άκρος ολοκληρωμένη η προσέγγιση. Διότι φαντάζεται σε μία κάποια προθεσμία που αναφέρεται 5 με 10% του προϋπολογισμού του ΑΕΠ να πηγαίνει στους προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής με το σεβασμό της δημοσιονομικής ουδετερότητας που είναι κάτι πολύ ουσιαστικό κυρίως έναντι των ε, πολιτών μας. Για τη συμβαστική 58 εκεί αναφέρεται ο κοινωνικός διάλογος στον μακροοικονομικό τομέα και ζητείτε μια ενίσχυση του ρόλου αυτού του διαλόγου. Έχουμε δύο τροπολογίες, δύο παραγράφους στα συμπεράσματα, ούτως πίν. Η πρώτη είναι η παράγραφος 59, η συμβιβαστική. Εκεί ζητείτε ξεχωριστή ψηφοφορία, έτοιμα του ΕΛΚ. Ίσως εκεί όμως έχουμε εξελίξεις. Έχουμε ένα αίτημα ξεχωριστή ψηφοφορία. όσον αφορά την ψηφοφορία με ειδική ψηφοφορία για την βάση για την φορολόγηση των επιχειρήσεων. Αυτό δημιουργεί πρόβλημα για το ΕΛΚ όσον αφορά την παράγραφο 59α νέα. Εκεί δεν υπάρχει υποστήριξη από την ομάδα ECR. Αυτή η παράγραφος ζητά ενδεχομένως εξελίξεις όσον αφορά την οικονομική διακυβέρνηση και αυτές οι εξελίξεις να μεταφράζονται μέσω μιας αναθεωρήσεως των συνθήκων και να γίνεται σεβαστή η κοινοτική μέθοδος. Αυτή είναι η τροπολογία του ΕΛΚ που πιστεύω ότι είναι σημαντικότατη. Εν συνεχεία, η δεύτερη παράγραφος των συμπερασμάτων είναι η 59 Β νέα. Εκεί μετά την τελευταία μας ε, συνάντηση, έκτοτε λοιπόν, Α, όχι, δεν είναι παράγραφο συμπερασμάτων, διορθώνει Μιλήτρια. Είναι... Ναι, είναι παράγραφο συμπερασμάτων. Λοιπόν, έγιναν και γίνονται διαπραγματεύσεις όσον αφορά το πώς θα εισαγάγουμε το σύμφωνο Europlus και από ό,τι κατάλαβα το ΕΛΚ μπόρεσε να δεχτεί μία από τις διατυπώσεις που είχα προτείνει, αυτή που εμφανίζεται στο κείμενό μας και που λέει ότι είναι πρωτοβουλία αυτό το σύμφωνο, μια πρωτοβουλία του Συμβουλίου. Στην παράγραφο 62, αλφανέα μάλλον, Εκεί ζητείται ξεχωριστή ψηφοφορία από πλευράς του ΕΛΚ με μια εναλλακτική πρόταση των σοσιαλιστών και δημοκρατών αλλά θα αφήσω την κάθε ομάδα να δικαιολογήσει την ξεχωριστή προσέγγιση που επιθυμεί διότι είναι η παράγραφος που δίνει μια γενική εικόνα, γενική προσέγγιση στα συμπεράσματα της εκθέσεως. Ζητώ συγγνώμη κύριε Πρόεδρε για αυτή την παρουσίαση που ήταν κουραστική, πολύ κουραστική, αλλά λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες εργασίας, θεώρησα σημαντικό κάποια από τα παρόντα μέλη να μπορέσουν να μπουν, να δουν αυτές τις λεπτομέρειες των υπραγματεύσεων. Ευχαριστούμε Πεχβάους. Θέλω να προτείνω το εξή. Έχουμε τις θέσεις όλων των πολιτικών ομάδων. Το ECR και το EFT πολύ συχνά έχουν διαφορετική άποψη. Αλλά δεν εκπροσωπούνται. Άρα δεν μπορούμε να το συζητήσουμε μαζί τους εδώ. Προτείνω τα σημεία στα οποία το ECR και το EFT θέλουν χωριστή ψηφοφορία ή θέλουν κάποια διαφορετική πρόταση, να το συζητήσουμε, να ψηφίσουμε αντίστοιχα τη Δευτέρα. Να τα αφήσουμε εντελώ δηλαδή αυτά τα θέματα. Δεν χρειάζεται καν να τα συζητήσουμε αφού δεν εκπροσωπούνται να ψηφίσουμε τη Δευτέρα για τα θέματα αυτά όπως το επιθυμούν. Στα άλλα σημεία στα οποία υπάρχουν διαφορετικές απόψεις και ζητούνται χωριστές ψηφοφορίες, αλλά από ομάδες που εκπροσωπούνται, δηλαδή ΕΛΚ, ε, Φιλελεύθεροι, ΓΚΟΕ και ε, Σοσιαλιστές και Δημοκράτες, να υποφεληθούμε της ευκαιρίας ε, από τους εκπροσώπους, δηλαδή από την παρουσία των εκπροσώπων ε, αυτών των πολιτικών ομάδων για να μας πούν αν μπορούν αυτά τα επίμαχα σημεία να τα διαγράψουν ή τέλος πάντων να δώσουμε κάποια λύση ή διαφορετικά θα πρέπει να ψηφίσουμε τη Δευτέρα για τα σημεία αυτά. Και να δώσω το λόγο στον Ότμαν, Ότμαν ε, Κάρας. Ο κύριος Η ΣΥΡΠΑ δεν ξέρω ποιος θα λάβει το λόγο να μας πει σε ποια σημεία ε, θέλει το ΕΛΚ χωριστή ψηφοφορία. Ή μήπως θέλετε κάτι να αλλάξουμε σε αυτά που έχετε προτείνει. Ο κύριος Κάρας. Κύριε Πρόεδρε, καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συνεργάτες ε, και όλων των ομάδων που δούλευσαν με όλους τους συναδέλφους για να μπορέσουμε να φτάσουμε στο σημερινό αποτέλεσμα. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται να ερμηνεύσουμε τώρα το ποιος έχει κάνει τι και γιατί. Υπάρχουν ε, πολλά σημεία στα οποία αν αρχίσουμε να τα συζητάμε θα διαφωνήσουμε και δεν υπάρχει κανένας λόγος ε, να μπούμε σε τέτοιες συζητήσεις. Νομίζω ότι ε, υπήρχε μια γραμμή στις συζητήσεις που δεν τροποποιήθηκε. Υπάρχουν λίγα σημεία στα οποία θα ήθελα να κάνω παρατηρήσεις. Το 7α ναι, το 19 ναι, στο 21 θα μπορούσαμε να κάνουμε και προφορική τροπολογία. Στο 21 πολλοί από εμά έχουν δυσκολία με τις λέξεις Economic Council, Οικονομικό Συμβούλιο. Το θέμα είναι αν μπορούμε να βρούμε ε, κάποια διαφορετική, κάποια εναλλακτική λύση ε, όσον αφορά την οικονομική διακυβέρνηση στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών. Γιατί δεν ξέρουμε τι κρύβεται πίσω από μια τέτοια έννοια που αναφέρεται εδώ. Αυτά όσον αφορά το Παγκόσμιο Οικονομικό Συμβούλιο και την Παγκόσμια Οικονομική Διακυβέρνηση στο πλαίσιο του Συστήματος των Ηνωμένων Εθνών. Ε, στο 27 μπορούμε να δεχτούμε αυτό το οποίο προτάθηκε το νέο. Στο σημείο essential παραμένουμε στη χωριστή ψηφοφορία. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται όμως να δικαιολογήσω τίποτα παραπάνω. Για το 37 σας ανέφερε η Περβόνς. Στο 38 πρέπει να πω ότι Δεν μιλάμε για δυνάμωση της ε, κατανομής κεφαλαίου. Και δεν νομίζω ότι εδώ ε, ε, μπορεί να μας βοηθήσει αυτό το οποίο αναφέρεται για, αναφέρθηκε για τα χρηματιστήρια. Το πρόβλημα τίθεται από τους όρους ε, dedicated stock exchanges. Και σε αυτό το σημείο ε, έχουμε ζητήσει την χωριστή ψηφοφορία. Για τα θέματα της εναρμόνισης και του συντονισμού έχουμε συζητήσει πολλές φορές Και εγώ συμφωνώ ε, να ε, συζητήσουμε τα θέματα που αφορούν τη φορολογία. Αλλά σε πολλές περιπτώσεις ε, μπορεί να τίθεται πρόβλημα από την παράταση μιας τέτοιας υποχρέωσης. Στο 40 νομίζω ότι μπορούμε να ψηφίσουμε έτσι ως έχει, γιατί νομίζω ότι μπορεί να υπάρξει συνένεση. Το 40 δεν θα θέλαμε ε, να μπει στην ε, ψηφοφορία μαζί με το 41. Έχουν γίνει πολλές συζητήσεις και σε εμά και σε άλλες ομάδες σχετικά με την αύξηση του προϋπολογισμού και αν θα έπρεπε να βάλουμε κάποιο, κάποιον αριθμό, να πούμε μέχρι 10%. Όσο σαφέστεροι είμαστε και όσο πιο ξεκάθαρη είναι η διατύπωση, τόσο το καλύτερο. Ελπίζω να υπάρξει υποστήριξη αν γίνει χωριστή ψηφοφορία ε, σε αυτά τα οποία αναφέρονται στην παράγραφο 57 για συγκεκριμένο αριθμό. Και ένα τελευταίο σημείο. Νομίζω ότι η έκθεση είναι καλύτερη σε σχέση με την προηγούμενη προσπάθειά μας, γιατί νομίζω ότι έχουμε γίνει πολύ πιο συγκεκριμένοι. Η πλειοψηφία στη δική μας ομάδα προτιμά να διαγραφούν κάποια επίμαχα σημεία αντί να τροποποιηθούν. Θέλουμε να έχουμε πιο ξεκάθαρη διατύπωση και οι τρεις συμπληρώσεις ε, τις οποίες ανέφερε η συνάδελφος ε, κυρία Μπερές ε, είναι τα σημεία στα οποία πιστεύουμε ότι πρέπει να είναι πιο ξεκάθαρα για να μπορέσουμε να έχουμε πλειοψηφία. Αλλά δεν θέλουμε ε, να υπάρξει πόλωση. Ε, μέχρι αύριο το μεσημέρι στις 12 ε, θα μπορέσουμε να δούμε τι περαιτέρω τροπολογίες μπορούν να υπάρχουν, ούτω ώστε μέχρι τη Δευτέρα να είναι σαφής η κατάσταση για την ψηφοφορία. Για το σημείο, για την τροπολογία 41 και για τις εναλλακτικέ στο πλαίσιο ε, του G20, είναι, ε, πιστεύω, οι δύο, τροποποιήσεις, οι δύο συμπληρώσεις οι οποίες μπορούν να γίνουν αυτή τη στιγμή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρο. Από ό,τι είπαμε στο Προεδρείο, ο κατάλογο ψηφοφορία θα σταλεί σήμερα μετά τη συνεδρίαση, οπότε μπορεί κάθε ομάδα να λάβει γνώση αυτή τη πρόταση και να σκεφτεί τον κατάλογο για την ψηφοφορία και μέχρι αύριο το μεσημέρι να μας ε, πει τη γνώμη του για το τι πιστεύετε ότι πρέπει να γίνει. Ένα σημείο, Ότμαρ, τώρα για το θέμα του προϋπολογισμού και για τον αριθμό το 5-10%. Ε, προσωπικά εγώ πιστεύω ότι εδώ προσπαθούμε να ψηφίσουμε, να διατυπώσουμε ε, την έκθεση όπως και στην Επιτροπή ΣΥΟΡ. Δηλαδή δεν θέλουμε να κάνουμε κάτι το οποίο θα βρίσκεται σε αντιπαράθεση με αυτό το οποίο θα ψηφίσει η Επιτροπή ΣΥΟΡ. Ο κ. Κάρας. Θα ήθελα να πω ότι αυτοί οι οποίοι πρότειναν εδώ τον αριθμό το συγκεκριμένο ε, δεν τον πρότειναν ε, και στη ΣΟΥΡ ε, γιατί νόμιζα ότι θα γίνει εδώ η ψηφοφορία, ότι θα ψηφίσουμε εδώ υπέρ της συμβαστική λύσης και όχι στη ΣΟΥΡ. Και ο προϋπολογισμός και οι προοπτικές, οι πολιτικές προοπτικές εδώ στη δική μας επιτροπή είναι πολύ πιο έντονες. Γι' αυτό υπήρξε ένα είδος συμφωνίας Ισου. Ε, Θα είναι αρμόδια για θέματα προϋπολογισμού. ούτως ώστε να μην δημιουργούμε προαπαιτούμενα και αυτά τα οποία κάνουμε εμείς εδώ να ε, ε, βοηθήσουν και τις συζητήσεις στη ΣΟΥΡ. Δηλαδή να ξέρουν και στην ε, ΣΟΥΡ ότι εμείς εδώ θα ασχοληθούμε με αυτή τη μακροπρόθεσμη προοπτική. Ευχαριστώ. Όλο Σμιτ. Ή, συγγνώμη. Σέτζο. Αλλά νόμιζα ότι η Περβόνς είχε Περβόνση ειχε μιλησει για, την μέρους των σοσιαλδημοκρατών. Ευχαριστώ. Κανένα πρόβλημα. Όμως, αναφερόμενος στις παρατηρήσεις που έκανε ο συνάδελφος Καράς, κάνοντας κάποιες σκέψεις πάνω σε αυτά, θεωρώ ότι η συμβαστική πρόταση που, στην οποία καταλήξαμε στην τελευταία συζήτηση, Οι προτάσεις είναι πολύ λογικές και αποτελεσματικές. Δεν βλέπω από πού γεννώνται κάποιες από τις ανησυχίες που ανέφερε ρητά ο συνάδελφος μόλις τώρα. Στο τέλος θεωρώ εξάλλου ότι υπάρχουν και άλλες παρατηρήσεις και επιληθέντα σημεία. Τα βασικά θέματα παραμένουν, στείνουν είναι τα θέματα τα σχετικά με τη φορολογική πολιτική. Όσον αφορά την παράγραφο 41, να υπενθυμίσω σε όλους σας ότι είχαμε βρει ένα είδος ισορροπίας δεν θέλω να το αποκαλέσω συμβιβασμό, αλλά μια ισορροπία προφανή. Ισορροπία μεταξύ του συντονισμού και της εναρμόνισης. Έγινε μακρά διαμάχη ανάλογα με το πώς οι διάφορες χώρες βλέπουν αυτά τα θέματα και τη διαμόρφωση μιας κοινής φορολογητές βάσης που κανείς δεν αφισβητούσε. Απ' την άλλη πλευρά καταλαβαίνει κανείς ότι αυτό είναι λογικό να συμβαίνει, διότι αν θέλει κανείς να εναρμονίσει ένα κοινό σημείο πρέπει να το έχει, αλλιώς δεν ξέρει από πού να ξεκινήσει και τι εναρμονίζει. Διότι εναλλακτική μιας βάσος όπως αυτή που έχουμε, όπως φανταστήκαμε για την παράγραφο 41, είναι να κάνουμε όλοι τα ίδια πράγματα. Δηλαδή, θα ήταν το ιδεώδες αυτό σε μια Ευρώπη εντελώς, τελείως ολοκληρωμένη. Όμως είναι, δεν είναι τόσο ραλιστικό το φανταστούμε σήμερα. Αν αλλάξουμε την ισορροπία αυτή, ανοίγουμε μια συζήτηση μεταξύ μας, η οποία ίσως δεν έχει λόγο ύπαρξης. Ο συντανισμός και η εναρμόνιση θα χρειαζόταν ένα κοινό σημείο που αυτή, αυτό το κοινό σημείο είναι η φορολογητέα βάση, κοινή βάση. Δεν βλέπω ανησυχίες όσον αφορά την προσέγγιση εγώ. Το δεύτερο θέμα τώρα αφορά τον προϋπολογισμό στις προηγούμενες συζητήσεις. Εμείς ενοποιήσαμε επιχειρήματα και θέματα που ήταν απομακρυσμένα, διάσπαρτα, ζητήματα που ήταν διάσπαρτα στην έκθεση. Και το κάναμε αυτό για να διασυνδέσουμε χωρίς να τα φέρνουμε σε αντίθεση αυτές τις δράσεις, αυτά τα σημεία όσα έπρεπε να γίνουν όσον αφορά τον προϋπολογισμό εγώ δεν πιστεύω στην αποτελεσματικότητα της χρήσεως των επιθέτων. Μία ποσοτικοποίηση είναι πολύ πιο περιοριστική από μία ένδειξη βούλησης, έκφραση βούλησης. Εδώ μιλάμε για μακροπρόθεσμους στόχους, όπως επανειλημμένα επενθύμησε η Περβάνς. Δεν είναι κάτι που ζητάμε να γίνει ε, μέσα σε μερικούς μήνες. Εάν βάλουμε της αναφοράς, όχι μόνο κάνουμε κάτι σωστό και συνεκτικό στο τέλος των εργασιών μας, αλλά κατά την άποψή μου έχουμε και την ευκαιρία να δώσουμε θετική όθηση συζήτηση που λαμβάνει η χώρα και σε άλλες επιτροπές. Γι' αυτό το λόγο πιστεύω ότι είναι χρησιμότατο να είμαστε στεναροί όσον αφορά την αναφορά των αριθμών. Διότι όπως έλεγα δεν έχει άμεση συνέπεια αυτό. Είναι μια πολιτική προπτικής. Να πω κάτι τελευταίο όσον αφορά τα, τις παραγράφους των συμπερασμάτων. Ε, τα σημεία παρέμειναν ανοιχτά. Ε, επιβεβαιώνω εκ νέου το ενδιαφέρον των σοσιαλιστών και δημοκρατών να έχουμε λύσεις που εντοπίστηκαν και ως συμβαστικές λύσεις, διότι μία έκθεση έχει συμπέρασμα συνοπτικό που συνοψίζει θέματα και επιχειρήματα που παρετέθησαν προηγουμένως. Λαμβάνω υπόψη ότι συνοψίζοντας μπορεί κανείς πάντα να παράγει, να πιέσει κάπως τα πράγματα, να μην βγει τόσο καλό. Συζητήσαμε όμως επί μακρόν στην τελευταία περίσταση τα λόγια, τις λέξεις που ε, ε, χαρακτηρίζουν τα διάφορα κεφάλαια. Εγώ νομίζω ότι είναι απαραίτητο να κλείσουμε την έκθεση με αυτή τη σύνοψη, τη σύνθεση που είναι συνεκτική και ταιριάζει με τη δουλειά εξάλλου που έγινε για την ε, έκθεση την ενδιάμεση. Διότι το σημαντικό είναι να έχουμε ένα συμπέρασμα το οποίο, ένα αποτέλεσμα που είναι η φυσική εξέλιξη στο βαθμό του δυνατού της προσέγγισης που ακολουθήθηκε στην ενδιάμεση έκθεση αλλά να μην αλλάζει τα, ε, τα διαβασικά στοιχεία και τους ευαίσθητους ε, συμβιβασμούς που εξευρέθησαν. Τόσο αναφορά αφορά τις λεπτομέρειες. Κανείς δεν αμφισβητεί ότι θα αφήσουμε για πάντα ανοιχτό το θέμα, γιατί διαφορετικά αμφισβητούμε και την αποτελεσματικότητα των συμβιβασμών και τα θετικά αποτελέσματα που υπελέγησαν αν εξακολουθούμε να παρατείνουμε τις εργασίες επαοριστών. Ε, Ευχαριστώ και τώρα θα δώσω το λόγο στον Όλε Σμιτ. Αλλά πριν αρχίσεις ε, Όλε, θέλω να ζητήσω για άλλη μια φορά συγγνώμη που πρέπει να φύγω. Δυστυχώς δεν έχουμε αντιπρόεδρο σήμερα, κανένα αντιπρόεδρο. Δεν έχουμε και κανέναν ουδέτερο που να μην είναι ούτε σκιώδης ούτε ε, συντονιστής. και οι συνάδελφοι θα μπορούσαν να είναι, δεν είναι εδώ. Όλε και μετά ο κ. Χουντής. <clears throat> Ευχαριστώ πολύ. Καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω την εισηγήτρια γιατί έχει κάνει πάρα πολύ δουλειά και πολύ αποτελεσματική. Και ευχαριστώ και όλους τους άλλους και τη γραμματεία και όλα τα μέλη του προσωπικού που μας βοήθησαν. Όπως πάντοτε στην πολιτική, κάποιος θα πρέπει να κάνει τη δουλειά για να μπορούμε εμείς να είμαστε πολιτικοί. Θα ξεκινήσω με ένα γλωσσικό σημείο, γιατί οι σπουδέ μου είχαν γλωσσικό περιεχόμενο και όλα πάλι με έλεγε πάντοτε ότι οι λέξεις σημαίνουν πολλά. Λέτε διαφάνεια και, αμοιβαίως, ε, και αμοιβαιότητα. Αυτό σημαίνει στην παράγραφο 13. Ε, αυτό σημαίνει ε, και χώρες ε, εκτό Ρωσίας και εκτός Ευρώπης, συγγνώμη, όπω η Ρωσία. Και μετά υπάρχει η λέξη balanced, ισορροπημένο, αλλά αν δεν σημαίνει δίκαιο εμπόριο, πάλι δεν θα με βρει σύμφωνο αυτή η λέξη. Μετά στην παράγραφο 41, έχουμε κάτι το οποίο είναι πολύ βασικό. Δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη του ΕΛΚ, αλλά εμείς θα θέλαμε να έχουμε ελεύθερο, ελεύθερο corporate tax base, την βάση επιβολή του εταιρικού φόρου να είναι ελεύθερη. Και σε κάποιες τροπολογίες των φιλελευθέρων αντικατοπτρίζεται αυτή η στάση. Θα προτιμούσα να καταλήγαμε όμως σε ένα κοινό κείμενο εδώ. Γιατί νομίζω ότι η τωρινή πρόταση του Επιτρόπου Σεμέτα αποτελεί ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Μετά για την 57... Άκουσα ότι η Σουέρ ακόμη διαπραγματεύεται τη συμφωνία. Και όπως έχω ξαναπεί, πιστεύω ότι αυτό το 5-10% δεν πρέπει να το έχουμε στο κείμενο διότι στην παρούσα κατάσταση των πραγμάτων δεν είναι αποδεκτό για τους πολίτες της Ευρώπης, οι οποίοι πρέπει να πληρώσουν. Καταλαβαίνω τη λογική ότι αν δώσουμε περισσότερα χρήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, θα πληρώνουν οι πολίτες λιγότερο σε εθνικό επίπεδο. Αλλά δεν ξέρω αν όντως θα συμβεί αυτό στην πράξη. Δεν είμαι βέβαιος. Πρέπει να υπάρχει συνέπεια σε όλο το κείμενο και σίγουρα θα το συζητήσουμε στην ομάδα μας. Εγώ θα προτιμούσα να λέμε adequate. Ο προϋπολογισμός θα πρέπει να είναι επαρκής. Έχω προβλήματα με το κείμενο. Εγώ, εγώ έχω προβλήματα με το κείμενο. Πρέπει να τονίσω το εγώ. Δεν ξέρω ο πρόεδρος αν έχει προβλήματα. Μετά στο 59... Φανήκατε πάρα πολύ έξυπνοι, κυρία Μπερές, γιατί έχουμε και πολλές τροπολογίες ε, των φιλελευθέρων, ακόμη και του επικεφαλής της ομάδας. Αυτό νομίζω ότι θα χρειαστεί να το μελετήσουμε λίγο. Νομίζω ότι θα είχαμε κάποιο συμβαστικό κείμενο σε σχέση με τα ευρωομόλογα. Τα ευρωομόλογα νομίζω περίπου μια εβδομάδα τα συζητάμε. Τουλάχιστον τρεις μέρες οπωσδήποτε. 48 ώρες. Δεν είμαι βέβαιος ότι θα λυθούν τα προβλήματα της Ευρώπης με αυτό. Πάντως εγώ θα ήθελα να έχουμε τα ευρωομόλογα στο κείμενο για την ε, οικονομική διακυβέρνηση. Στην ομάδα μας ε, είχαμε ένα κανόνα τον οποίο ακολουθήσαμε σε σχέση με το κείμενο. Αλλά θα πρέπει να ξαναρωτήσω. Δεν ξέρω αν ε, ο πρόεδρος ε, το θεωρεί αποδεκτό αυτό ως έχει. Μετά έχουμε το 62α νέο. Και θα ήθελα να ρωτήσω αυτούς που συνέταξαν το κείμενο, χωρίς να θέλω να φανώ αγενής. Ε, τι είναι το νέο που έχουμε εδώ. Τι είναι αυτό το New European Deal που έχουμε εδώ. Το Ρούσβελτ μου θυμίζει αυτό. Νομίζω ότι κάπως θα έπρεπε να το αναδιατυπώσουμε. Μου φαίνεται υπερβολικό. Δεν ξέρω πώς ακριβώς να το πω, αλλά για να το καταλάβω και για να μπορέσω να, να το δεχτώ χρειάζομαι κάποιες επιπλέον εξηγήσει. Ευχαριστώ. Ο κύριος Χουντής, πρώτο ο ομιλητής και Χανσπέτερ Peter Μάρτιν, αλλά πρώτο ο κύριος Χουντής. Ε, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Στις εκκρεμότητες που έχουν μείνει σχετικά με τους συμβιβασμούς δεν έχω να προσθέσω τίποτα καθώς οι συμβιβαστικές προτάσεις που έχουν μείνει με κάποιες εκκρεμότητες ε, δεν αφορούν τροπολογίες τις οποίες έχουμε καταθέσει εμείς. Με αυτή την έννοια, σε αυτή τη διαδικασία είμαστε ουδέτεροι και επειδή φεύγει ο Πρόεδρος προσφέρομαι να, αν δεν υπάρχει αντίρρηση να, συνε... να προεδρεύσω την έννοια της ουδετερότητας. <laughs> Ναι, ναι. I'm joking. I'm joking. <laughs> Ωραία. Ε, <laughs> ωραία. Λοιπόν, ε, θέλω ε, να πω δύο λόγια ακόμα. Θέλω να πω δύο λόγια ακόμα. Ε, έχω εξηγήσει γιατί το κείμενο δεν μας βρίσκει σύμφωνους, παρά το σεβασμό στην προσπάθεια που έχει γίνει. Θα δούμε τις τροπολογίες, αναφέρονται ήδη στο κείμενο, κάποιες που λαμβάνουν υπόψη και τις δικές μας παρατηρήσεις και αντίστοιχα θα τοποθετηθούμε σε αυτές τις τροπολογίες. Ε, τρίτο, Θέλω να αναφερθώ στην προσθήκη που μας προτείνει σήμερα η εισηγήτρια σχετικά το να μπει στο σκεπτικό μια αναφορά με το Σέγγεν. Ναι, θέλω να κάνω μια αναφορά. Μέχρι που να πάω στην τελευταία πρόταση δεν καταλάβαινα γιατί μια αναφορά για το Σέγγεν και τις εξελίξεις πρέπει να μπει στο δικό μας κείμενο. Μέχρι που να πάω στην τελευταία πρόταση της ε, τροπολογίας που μας δώσατε, της προσθήκης αν κατάλαβα όμως διαβάζοντας την τελευταία πρόταση, δεν ξέρω αν αυτό, επιτρέψτε μου να πω, αυτός ο εκβιασμός, προσέξτε, αν περιοριστεί η ελευθερία στη μετακίνηση των προσώπων, αυτό σημαίνει απειλή και στη μετακίνηση του κεφαλαίου, προς τα πού απευθύνεται και πώς μπαίνει στο δικό μας το κείμενο. Εν πάση περιπτώσει, αυτή είναι μια επιφύλαξή μου. Κατά τα άλλα, επί της ουσίας, για τις μονομερείς αλλαγές και τα μέτρα που παίρνονται από ορισμένε χώρε προφανώ δεν συμφωνούμε. Δεν θέλω να σα κουράσω περισσότερο παρά μόνο λέγοντα ότι εκτιμώντα και σεβόμενο την προσπάθεια που έγινε όλο αυτό το διάστημα και τη συζητήτρια και των άλλων σκιωδών και από εκτίμηση και σεβασμό με τη συνεχή μα παρουσία προσπαθήσαμε να, να πείσουμε για ορισμένα πράγματα, δεν τα καταφέραμε. Επομένω ε, τη Δευτέρα θα είμαστε μαζί στη φωτογραφία αλλά στην ψηφοφορία θα ψηφίσουμε διαφορετικά. Μαζί στη φωτογραφία λόγω της κοινή προσπάθειας και του σεβασμού και της εκτίμησης, αλλά δεν θα την ψηφίσουμε την έκθεση. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ. Επιθυμεί κάποιος άλλος να πάρει το λόγο. Ο κ. Hans Peter Martin. Äh, ευχαριστώ, Πρόεδρε για λόγους υγείας ε, δεν μπόρεσα να συνεργαστώ μαζί σας στο βαθμό που θα το επιθυμούσα. Τη διαδικασία τη θεωρώ πολύ ενδιαφέρουσα. Είναι κρίμα που ε, δεν έτυχε μεγαλύτερη προσοχή και δημοσιότητα ε, η δουλειά τη Επιτροπή. Και αν ήταν και ο Πρόεδρο εδώ, θα τον ρωτούσα μετά από 1,5 χρόνο, κατά τη γνώμη του, ποια είναι η προστιθέμενη αξία πέραν της διαδικασίας. Δηλαδή, κατά τη γνώμη του Προέδρου, τι είναι αυτό που μπορούμε να πούμε ότι προσφέρουμε στους πολίτες. Δεν είναι όμως εδώ ο Πρόεδρος. Ίσως θα μπορούσε η συγγήτρια ε, εν συντομία να μου απαντήσει. Ευχαριστώ. Μήπως επιθυμεί κάποιος άλλος να πάρει το λόγο. Δεν μου φαίνεται. Να σας ευχαριστήσω για μία ακόμη φορά. Ευχαριστώ, Hans Peter Martin, για την ερώτησή σας, διότι με τα χαράς θα απαντήσω σε αυτήν στο τέλος της ε, συζητήσεως. Πριν το κάνω αυτό, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους για αυτά που είπαν και ίσως θα ήθελα να επανέλθω σε ένα-δύο σχόλια του συναδέλφου Όλε Σμιτ, διότι αυτές οι παρατηρήσεις αφορούσαν τα πιο συγκεκριμένα σημεία. Όσον αφορά την παράγραφο για την φύση των συναλλαγών, πράγματι θέλαμε δίπλα στο free trade να βάλουμε balanced and fair trade, ισορροπημένο και ελεύθερο εμπόριο αντί ελεύθερο εμπόριο. Αν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα στο παγκόσμιο εμπόριο που γνωρίσαμε, οι ελεύθερες συναλλαγέ δεν αρκούν. Ξέρω ότι είστε πολύ φιλελεύθερος, ότι είναι πολύ φιλελεύθερο αυτό, αλλά πέρα από την ελεύθε, τις ελεύθερες συναλλαγές, η ιδέα συναλλαγών ισορροπημένων και δικαίων θεωρώ ότι είναι κάτι πολύ σημαντικό και διαπιστώνω ότι στο συμβιβασμό που επεξεργαστήκαμε ε, υπάρχει μια συμφωνία κανονικά πάνω σε αυτό. Όσον αφορά τη φορολόγηση των εταιριών, την ενοποιημένη βάση, την ενιαία βάση. Στην Οικονομική Νομισματική Επιτροπή θα εξαχθεί συζήτηση όταν θα εξετάσουμε την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δεν θα πρέπει να, να προκαταλάβουμε εδώ τη συζήτηση που θα διεξαχθεί. εφόσον όμως είναι ανοιχτό το θέμα, παίζεται το εξή. Κατά πόσο θα πρέπει να είναι υποχρεωτική ή ε, εθελοντική η θελοντικη η εναρμονιση της βάσης. Ειλικρινά πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό θέμα αυτό. Πολύ σημαντική συζήτηση, διότι αν η εναρμόνιση, να το πω ειλικρινά, εάν αύριο κάνουμε μια εναρμόνιση της βάσης της φορολόγησης των εταιριών, επιδυνητικής βάσος, επιθελοντικής βάσος, αυτό δεν θα επιτρέψει ποτέ να ξαναοικοδομήσουμε τη φορολογική βάση των κρατών μελών. Θα επιτρέψουμε μόνο στις ε, πολυεθνικές να βελτιστοποιήσουν το, τη χώρα, τον τόπο της φορολόγησής τους. Νομίζω ότι εξάλλου θα το ψηφίσουμε. Ε, για την παράγραφο 57 και τη διαφορά αυτή που έχουμε τη διχάλα από 5 μέχρι 10%. Δεν θα επαναλάβω αυτά που μας είπε ο συνάδελφος ο κ. Κάρας, αλλά πολλά που συμπεριλαμβάνονται σε αυτή την έκθεση, όπως και στην προηγούμενη έκθεση, ε, δεν έχουν συντονιστεί απόλυτα. Ε, γνωρίζουμε τι τρέχει. Δεν ξέρουμε μάλλον τι τρέχει ούτε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ούτε στο Συμβούλιο. Σε αυτό το πνεύμα από την αρχή θεωρήσαμε ότι χρειάζεται κάποια στιγμή σε ευρωπαϊκή κλίμακα κάποιος, κάποια ομάδα να προβάλλει ένα πιο φιλόδοξο όραμα, ε, πιο μακροπροθέσμο όραμα που θα προστατεύει η Ευρώπη τους πολίτες εν μέσω παγκοσμιοποίησεως και σε, εντός των κρίσεων. Κανείς δεν θεωρεί ότι αύριο το πρωί θα φτάσουμε στο 5-10%. Ούτε καν στο τέλος της, στο τέλος της επομένης περίοδου των δημοσιονομικών προοπτικών. Αλλά ο στόχος υπάρχει να πούμε ότι χρειαζόμαστε μια ισχυρότερη, πιο ολοκληρωμένη Ευρώπη, άρα με τα μέσα να υπομειστεί τις ευθύνες της και στο παγκόσμιο επίπεδο και έναντι των πολιτών μας. Για μια ακόμη φορά να πω ότι ελπίζω ότι αγαπητοί συνάδελφοι θα μπορέσετε να εξηγήσετε εσείς οι ίδιοι στους πολίτες σας. Να μην τους πείτε ότι σήμερα, να τους πείτε σφίξτε το ζωνάρι σε εθνικό επίπεδο και σε ευρωπαϊκή κλίμακα να σπαταλάτε όλα αυτά τα χρήματα και να τα πετάτε στους γραφειοκράτες των Βρυξελών. Δεν είναι το πνεύμα αυτού που προτείνουμε. Αυτό που προτείνουμε είναι φορολογική ουδετερότητα για τους πολίτες. Αυτό αναφέρεται σαφώς στο παραγράφου και είναι μακροπρόθεσμη η προοπτική. Για να δείξουμε ποιο είναι το μονοπάτι. Να πούμε ότι αύριο όταν θα γίνουν οι διαπραγματεύσεις για δημοσιονομικές προοπτικές που θα είναι ένας εφιάλτης όπου οι Βρετανοί θα πολεμήσουν για τα χρήματά τους, για τους έκτους, οι Πολωνοί για την πολιτική συνοχή, η Γαλλία θα πολεμήσει για την αγροτική πολιτική, η Γερμανία θα πολεμήσει για να μην πληρώσει σεντ παραπάνω, ούτε ένα ευρώ παραπάνω για τον ευρωπαϊκό προπολογισμό, θα είναι ένας εφιάλτης. Εμείς λέμε ότι ξέρουμε πολύ καλά ότι ακόμα και αν σε επίπεδο συμβουλίου θα είναι φρικτές οι διαπραγματεύσεις, διότι είμαστε σε δύσκολο πλαίσιο, θα πρέπει η αρχή όμως να συμπεριλαμβάνεται για την 59 Συμμερίζομαι την ιδέα σας και υπενθυμίζω ότι ήδη στην πρώτη έκθεση είχαμε αναφερθεί στην προπτική των project bonds και του επιμερισμού των χρεών. Πιτικά είναι μας επέτρεψε να κάνουμε μια σωστότερη διατύπωση για την αμοιβαία έκδοση χρεογράφων. Λοιπόν, ήταν κάτι που αναφέραμε και στην πρώτη έκθεση και αναφέρθηκε και στο πακέτο για την οικονομική διακυβέρνηση. Σε αυτό το πλαίσιο της σύνοψης ελπίζω να μπορέσουμε να συμπεριλάβουμε σωστά την όρια διατύπωση. Όσον αφορά την 62α νέα, ίσως ανάμεσα στις ομάδες να εξακολουθεί να υπάρχει ε, κάποια διαφωνία. Θα δούμε πώς θα παρουσιαστεί ο κατάλογος των ψηφοφοριών τη Δευτέρα θα δούμε αν μπορούμε να συζητήσουμε ακόμα τα κείμενα σήμερα. Ε, αυτό η νέα συμφωνία New European Deal ε, δεν με ενοχλεί. Αυτή είναι η Ευρωπαϊκή Συμφωνία New European Deal διότι σαν παρατηρήτρια ή σαν συμμετέχουσα στην Ευρωπαϊκή Οικοδόμηση επί σειρά ετών νομίζω ότι τα μικρομαστορέματα που κάνουμε καθημερινά δεν μας εγγυώνται ότι θα ε, τα καταφέρουμε στο τέλος. Και οι συζητήσεις που έγιναν στο τελευταίο Συμβούλιο ΕΚΟΦΗΝ όσον αφορά την κατάσταση στην Ελλάδα μας το δείχνει αυτό. Υπάρχουν πολλά πράγματα που θα πρέπει να κάνουμε εμείς αν θέλουμε να είμαστε βέβαιοι ότι αυτός ο χώρος της αλληλεγγύης, της συγκλήσεως που οικοδομήσαμε μετά από πολλά χρόνια θα τα καταφέρει να βγει, όχι ζημιωμένο, να βγει και ε, ενισχυμένο, το οικοδόμημα από αυτή την κρίση. Λάβατε επίση μια πρόταση προστίκη, μια παραγράφο όσον αφορά το Σέγγεν. Ε, ε, δεν είναι μια παράγραφος που χαλάει την ισορροπία. Η αναφορά στο Σέγγεν δεν είναι καθόλου ουδέτερο όμω. Ο κύριος Χουντής μας εγκατέλειψε, έφυγε. Νομίζω ότι αυτό που λέει αυτή η τροπολογία είναι το εξή. Όταν εκατομμύρια Ευρωπαίοι έκαναν αυτό το σημαντικό βήμα στην ευρωπαϊκή οικοδόμηση, δηλαδή η δημιουργία του ευρώ, πάντα και ο Χέλμουτ Κόλ και ο Φρανσουά Μιτεράν πίστευαν ότι όλα αυτά μας οδηγούσαν σε μια πολιτική ένωση. Ήταν μια διαδικασία για να προχωρήσουμε πιο μακριά η δημιουργία της πολιτικής ένωσης, η ελεύθερη διακίνηση των ατόμων δεν είναι κάτι ίσονο σημασία, δεν είναι κάτι αμεληταίο. Εάν υπονομεύσουμε, λοιπόν, αμφισβητήσουμε την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων, η επιβίωση της Ευρωζώνης ίσως αμφισβητηθεί. Διότι δεν φαντάζομαι εγώ ένα χώρο όπου θα μπορούμε να δεχόμαστε την ελεύθερη διακίνηση των κεφαλαίων, υπαναχωρούμε στην ελεύθερη διακίνηση των ατόμων και η όλη ισχύ του εννοιαίου νομίσματος να μπορεί να επιβιώσει. Αυτό είναι το μήνυμα που βγαίνει από εδώ. Αυτό προτείνω να συμπεριλάβουμε αυτή την παράγραφο που αναφέρεται στο Σέγγεν. Και είμαι έτοιμη να το, να το αντιτυπώσουμε. Όσον αφορά αυτό που είπε ο κ. Hans Peter Μάρτιν, ευχαριστώ που θέσατε το ερώτημα. Καταρχάς δεν εργαστήκαμε τον ίδιο τρόπο στην πρώτη και τη δεύτερη φάση. Διαπιστώνω επίσης βλέποντας τι πετύχαμε σε αυτό το κοινοβούλιο πιστεύω ότι υπήρχε το μήνυμα που προανέφερα. Έβγαινε το μήνυμα, δηλαδή στην κρίση που αντιμετωπίζουμε σήμερα υπάρχει ένα θεσμικό όργανο όπου τολμούμε να, τολμά να σκέφτεται ότι υπάρχει ένα μέλλον φιλόδοξο για την Ευρώπη. Δεν είναι πάντα της μόδας να υπερασπίζεται σήμερα κανείς την Ευρώπη. Αλλά πιστεύω ότι είναι σημαντικό οι πολιτικοί υπεύθυνοι να έχουν επίγνωση ότι μπορούν να αντισταθούν στον εθνικισμό, στον λαϊκισμό και να πούνε ναι το μονοπάτι στο οποίο ξεκινήσαμε μαζί να περπατάμε το 57 το μονοπάτι που πρέπει να ξεκούσουμε να περπατάμε και χρειάζεται μεγάλη αλληλεγγύη κινητοποίηση για να βγούμε από την κρίση. Σημερίζομαι εν μέρη τα ερωτηματικά σα στο εξή. Αν σε αυτή τη δεύτερη φάση των εργασιών μα, μήπω θα έπρεπε να έχουμε μεγαλύτερη συνένεση. Θέλαμε στη δεύτερη φάση να έχουμε μεγαλύτερη συνένεση από ό,τι στην πρώτη. Και έτσι κινηθήκαμε. Μήπως μπορούσαμε να ακολουθούσαμε άλλη προσέγγιση. Να έχουμε μια Επιτροπή Έρευνας όσον αφορά το ελληνικό, πώς αντιμετωπίστηκε τις αγορές στο ελληνικό κρατικό χρέος και πώς παρενέβησαν οι επενδυτικές τράπεζες στις διάφορες αναπτυξιακές, στις φάσεις αναπτύξης αγοράς. Δεν κάναμε συλλογικά αυτή την επιλογή. Θα πρέπει αυτή η ειδική επιτροπή έπρεπε να ανοίξει το μονοπάτι σχετικά με το ευρωπαϊκό μέλλον. Αυτό πρέπει να το κάνουμε αν δεν θέλουμε να καταστρέψει αυτή η κρίση το όνειρο των ιδρυτών πατέρων. Δεν νομίζω να κάλυψα πλήρως ερωτήσεις σας και σας καλώ αν θέλετε να δείτε τη δουλειά που έκανε η Επιτροπή μας στην ισοσελίδα το έγγραφο που λέει ότι όλε οι προτάσει εκθέσεω τη Ειδική Επιτροπή που υφίστηκαν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν θα γίνουν πραγματικότητα παρά μόνο αν το Συμβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενστερνιστούν αυτέ τι προτάσει. Αυτή είναι η δουλειά των βουλευτών που εργάζονται σε μια ειδική επιτροπή που έγινε. Ευχαριστώ πολύ. Ε, σας απασχολήσαμε τις εργασίες μας σήμερα. Εν ονόματι του Προέδρου της Επιτροπής αυτής σας δίνω ραντεβού για την ψηφοφορία την Δευτέρα.